Συνάδελφοι, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε. Ναι, είναι η γνωστή παροιμία ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να περιμένουν αυτοί που ήρθαν στην ώρα τους. Και Εννοείται ότι δεν θα πρέπει αυτοί να τιμωρηθούν. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην τελευταία μας συνεδρίαση αυτής της περίοδου. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται με την παρούσα μορφή η ημερήσια διάταξη και μπορούμε να περάσουμε στα πρακτικά, τα σχέδια πρακτικών της 20ης ε, Φεβρουαρίου αλλά και της 11ης Μαρτίου υπάρχουν στους φακέλους σας. Έχετε κάποια σχόλια, παρατηρήσεις, όχι. Θα ήθελα αμέσως να σας προτείνω να θεωρήσουμε αυτά τα πρακτικά εγκεκριμένα, εκτός βεβαίως εάν υπάρξουν κάποια σχόλια κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης όσον αφορά την διερμηνία, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, τσεχικά, βουλγαρικά, ιστονικά και ρουμανικά. Σε αυτές τις γλώσσες παρέχεται η διερμηνία και βεβαίως θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή ακριβώς είναι η τελευταία μας συνεδρίαση, είναι απαραίτητο οι αποφάσεις, ιδιαίτερα των ε, συντονιστών της συνεδρίασης που μόλις έλαβε χώρα να σας ανακοινωθούν ε, προφορικά έτσι ώστε να είμαστε και τυπικά εντάξει. Οι αποφάσεις των συντονιστών είναι εξή πρώτον όσον αφορά οι τρεις αναφορές της Επιτροπής Αναφορών όσον αφορά την αντικειμενικότητα για την έκφραση απόψεων και τα μέσα ε, μαζικής ενημέρωσης έγιναν δεκτές και θα αποσταλούν στην Επιτροπή Αναφορών όσοι έχουν. Δεύτερον, όσον αφορά την γνωμοδότησή μας για τον προϋπολογισμό 2020, που υπομορφήν ε, επιστολής ε, θα αποσταλούν από την Πρόεδρο στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και αυτό εγκρίθηκε από τους συντονιστές. Επίσης, όσον αφορά τα προσυνημέρωση έγγραφα, Εκεί δεν υπήρξε, αν θέλετε, καμία απόφαση, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για περαιτέρω δράση, ενημερωθήκαμε. Αυτές είναι, νομίζω, οι αποφάσεις των συντονιστών, δεν νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες. Οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται οι αποφάσεις των συντονιστών της σημερινής συνεδρίασης. Την Τετάρτη την προηγούμενη Τετάρτη, συγγνώμη, ε, δημοσιεύθηκε η έκθεση που είχαμε ζητήσει για αυτούς που εγκαταλείπουν νωρίς στο σχολείο. Πρόκειται για ένα έγγραφο εξαιρετικό. Θα άξιζε τον κόπο να το κοιτάξετε με μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως ε, η επόμενη Επιτροπή Πολιτισμού σίγουρα θα συνεχίσετε την επεξεργασία αυτών των προτάσεων. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ σοβαρή δράση στην Ευρώπη γιατί είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολούσει. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι νέοι καταλείπουν πολύ νωρίς το σχολείο. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα της εμερήσης διάταξης που αφορά τις ψευδείς ειδήσει. Πρόκειται για την ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2019 οι συντονιστές της Επιτροπής μας πήραν την απόφαση να καλέσουν εκ νέου την Επιτροπή καθότι όλοι ξέρουμε ότι η η έκθεση της Επιτροπής, θέλουμε να μας τα την παρουσιάσει. Πρόκειται για την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ε, ειδήσει ε, στο διαδίκτυο εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η δημοκρατία, η σωστή λειτουργία της δημοκρατίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της ενημέρωσης των πληροφοριών που λαμβάνουν οι πολίτες μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό πώς μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα των πληροφοριών. Είναι μια βασική προϋπόθεση αυτή για να υπάρχει εμπιστοσύνη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και για όλους τους ε, θεσμούς πολιτικούς και επιστημονικούς. Πιστεύω ότι αυτή η κοινή διαπίστωση και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια συμφωνούμε όλοι ότι αυτά τα fake news, οι ψευδείς ειδήσει, η παραπληροφόρηση είναι ένα μαζικό φαινόμενο και μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί από πολιτικούς αντιπάλους για να πλήξουν την αξιοπιστία κάποιων θεσμών θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω θερμά τον Γενικό Διευθυντή Βιόλα της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Θα μας δώσει κάποια επιμέρους στοιχεία, θα μας παρουσιάσει την έκθεση και βεβαίως τον κώδικα ε, ορθής πρακτικής δεοντολογίας που υπάρχει μόνο στα αγγλικά από ό,τι ξέρω. Κοιτάξτε, το κείμενο συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και στη γερμανική ιστοσελίδα στα αγγλικά. Εγώ πιστεύω και δεν νομίζω ότι αυτό είναι μόνο δική μου άποψη. Όλοι οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν ότι τουλάχιστον αυτό το κείμενο είναι απαραίτητο να μεταφραστεί και να υπάρχει ε, σε ανάρτηση στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν να ενημερωθούν οι πολίτες της Ευρώπης για αυτόν τον κώδικα που αφορά ένα τόσο σοβαρό θέμα, την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσει. Νομίζω λοιπόν ότι για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα αυτό. Ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία δίνουμε στο να υπάρχουν αυτά τα σημαντικά ε, κείμενα σε όλες τις γλώσσες. Ναι, τα γαλλικά και τα αγγλικά μπορεί να είναι οι πιο διαδεδομένες γλώσσες στην Ευρώπη. Όμως, για ένα τέτοιο θέμα ε, μου είναι παντελώς ε, αδιανόητο να παραμείνουμε μόνο στην αγγλική γλώσσα. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, θα πρέπει αυτό να αλλάξει και να διορθωθεί αυτό το σφάλμα. Κύριε Βιόλα, σας καλωσορίζω και σας δίνω το λόγο για περίπου 10 λεπτά. Ε, πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε στην ε, συνεδρία της Επιτροπής σας. Είναι η τελευταία αυτής τη κοινοβουλευτική θητεία. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλους, όλα τα μέλη τη Επιτροπή για τη θαυμάσια δουλειά που κάνετε και για τη θαυμάσια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον υποφαινόμενο ιδιαίτερο. Για πολλά πράγματα συνεργαστήκαμε, πολλά επιτύχαμε. Θα ήθελα όμω να υπενθυμίσω τη μεταρρύθμιση των κανόνων για τα οπτικοακουστικά, την ε, οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες που είναι μια μοναδική νομοθεσία στον τομέα της. Ε, τη συζητήσαμε, ε, μιλήσαμε για τα νέα μέσα ενημέρωσης, ε, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και τα νέα πρότυπα για τη ρυθμίσή τους. Σας ευχαριστώ για αυτή τη σημαντική δουλειά, για το σημαντικό αυτό έργο και για την η οθέτηση αυτή τη σημαντική νομοθεσία. Σήμερα συζητάμε για τι ψευδεί ειδήσει, την παραπληροφόρηση και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπω είπατε, για το μέλλον τη Ευρώπη και ιδίω για τι επερχόμενε ευρωπαϊκέ εκλογέ. Σε μια απόπειρα να προσδιορίσω τι είναι τα ψευδή νέα πρέπει να πω ότι βέβαια δεν είναι εύκολο. Ε, ας μιλήσω για το φάσμα των ψευδών ειδήσεων. Ποιο είναι αυτό το φάσμα. Ξεκινάμε από τις κοινωνικές, κοινωνικά διαμορφωμένες επιθέσεις α, που είναι μία απόπειρα ενός κράτους ή ιδιωτικό φορέα να αποσταθεροποιήσουν μία κρατική οντότητα ή μία κοινωνική ομάδα. Υπάρχει σαφής πρόθεση και Υπάρχει απόπειρα προσβολής της ε, δημοκρατικής ε, τάξης, δημιουργίας πανικού ή οτιδήποτε άλλου, άλλου προβλήματος. Αυτό είναι κυβερνοεπιθέσει. Ε, σε ό,τι αφορά, τι πούμε, τις ελεύθερες εκλογές που γίνονται σε πολλά κράτη, αυτό είναι και έγκλημα. Από εκεί, λοιπόν, φτάμε σε επιθέσεις που δεν είναι προσδιορισμένες χρησιμοποιούνται απλώς τα κοινωνικά μέσα για να δημιουργηθεί πανικός, ε, συναισθήματα ε, με την εξάπλωση πληροφοριών που, κοινωνικά, που προκαλούν κοινωνική αποσταθεροποίηση ή αλλάζουν την ε, δημόσια τάξη στην κοινωνία. Παραδείγματο χάρη ψευδεί ιατρικέ ειδήσει. Τι επιπτώσει θα μπορούσαν να έχουν και τι απειλή συνιστούν για το ευρωπαϊκό σύστημα υγείας. Εν συνεχεία, έχουμε έναν άλλο τομέα όπου είναι ακόμα πιο περίπλοκο να κρίνουμε σε ποιο τομέα βρισκόμαστε. Ε, η δημιουργία απόψεων με τη χρήση στοιχείων που με βάση τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι σωστά, είναι βάσιμα για να αποκτήσει κανείς πολιτικό πλεονέκτημα και φτάνουμε στην άλλη πλευρά του φάσματος ε, που αφορούν το πολιτικό περιεχόμενο, την ε, ελευθεροτυπία, ε, την ορθότητα κτλ. Καταλαβαίνετε πόσο περίπλοκο λοιπόν είναι το θέμα από όλο αυτό το φάσμα. Ε, ξεκινάει από την κυβερνοασφάλεια ε, και φτάνουμε μέχρι θέματα ελευθερίας λόγου. Φυσικά υπάρχουν ψευδείς ειδήσει και υπήρχαν ψευδείς ειδήσει στην ιστορία, αλλά σήμερα είναι πολύ πιο σημαντικά, γιατί τα πραγματικά ε, κοινωνικά μέσα πολλαπλασιάζουν αυτή την αίσθηση, αυτό το συνέστημα του κόσμου. Ε, ο κόσμος νομίζει κάποια πράγματα ότι είναι άσχημα, ε, ότι είναι πάρα πολύ τρομακτικά. Υπήρχαν αυτά στην ιστορία, αλλά τα κοινωνικά μέσα παίζουν το ρόλο του πολλαπλασιαστή. Και αυτό είναι πολύ απλητικό. Οι νέε τεχνολογίες λοιπόν λειτουργούν πολλαπλασιαστικά λοιπόν, και δημιουργούν αυτή την κλίμακα του φαινομένου. Λόγω φύση λοιπόν, από νομικής άποψης, από τεχνικής άποψης, από κοινωνικής άποψης, ε, αντιμετωπίζουμε ένα πολύ περιπλοκό φαινόμενο. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να βρούμε μια εύκολη λύση για αυτό το πρόβλημα και θα χρειαστεί πολύς χρόνος πριν καταλάβουμε τα πάντα, πριν να ε, καταλάβουμε ας πούμε πώς αντιδρά Αυτά αυτό είναι το γενικό, το μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Θέλω να επανέλθω και στο βραχυπρόθεσμο πρόβλημα, τη εκλογέ. Έχουμε τη νέα οδηγία για τα οπτικοακουστικά. Υπάρχει ο σπόρο, α πούμε, για τη μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα, που είναι ε, γνώση του πώ λειτουργούν τα μέσα ενημέρωση. Έχουμε μια γενιά μαθητών που έχουν εκπαιδευτεί με την ιδέα ότι η ιστορία μπορεί να αναδιαμορφωθεί, να τη χειραγωγήσει κανείς. Τη μάθανε στο σχολείο ξανά και ξανά. Ή μάλλον, ε, κάποιοι μαθητές τη μάθαν στο σχολείο και είναι δεδομένοι. Αλλά κάποιοι άλλοι ε, μεγαλώνουν με τα κοινωνικά ε, μέσα ενημέρωση και μαθαίνουν την ιστορία μέσα από αυτά. Ε, Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξέρει κανείς από τα, να ξέρει κανείς από τα, μέσα, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, ε, γιατί είναι το πραγματικό εμβόλιο. Αυτή η νέα οδηγία έχει εισαγάγει την υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την ε, γνώση των μέσων ενημέρωσης και την υποχρέωση για τις πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων να προωθήσουν τη γνώση του πώς λειτουργούν δηλαδή αυτά τα μέσα ενημέρωσης πάμε στο βραχυπρόθεσμο πλαίσιο. Το Δεκέμβριο υιοθετήσαμε ένα σχέδιο δράσης και επανήλθαμε με ένα συμπληρωματικό πακέτο. Ξεκινήσαμε με μία διαβούλευση των ενδιαφερομένων ομάδων και το, πιο λογικό, το πρώτο λογικό ε, βήμα σε αυτό το δύσκολο ταξίδι είναι η αυτορύθμιση. Ε, ο ελεύθερος, η ελεύθερη έκφραση όμως ε, μπερδεύεται με πράγματα που έχουν κοινωνική σημασία. Ε, προσπαθούμε λοιπόν σε μια πρώτη φάση να ρυθμίσουμε το πρόβλημα με την αυτορύθμιση. Ζητάμε από τις πιο σημαντικές πλατφόρμες να έχουν ένα κώδικα αυτορύθμισης, ε, τον υιοθέτησαν αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη δέσμευση που πήραν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι δεσμεύσεις αποτελούνται από πολλά πράγματα. Το πιο σημαντικό, αυξάνεται ο έλεγχος σε ψευδείς λογαριασμούς, εξασφαλίζουν ότι προωθούνται οι έμπιστες πηγές και σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κόμματα ε, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, και αυτές είναι οι βασικές δεσμεύσεις. Αυτές οι δεσμεύσεις όμως πρέπει να πάρουν ας πούμε σάρκα και οστά. Γι' αυτό λοιπόν εν των εκλογών θα πρέπει ε, να μας ε, υποβάλουν εκθέσεις μηνιαία για να μας εξηγούν ποια είναι η πρόοδος. Υπάρχουν δύο εκθέσεις για την εφαρμογή αυτού του ε, κώδικα αυτορύθμισης και είπαμε δημοσία ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλοί τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Παραδείγματο χάρη, αύξηση της διαφάνειας στα πολιτικά θέματα, ε, προβλήματα με τους ε, ψευδείς ε, λογαριασμούς. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρότυπο όμως. Πώς μετράμε την επιτυχία σε αυτό το τομέα και πόσο γρήγορα και σοβαρά προωθούμε αυτό το έργο. Αλλά ως αφετηρία θεωρούμε ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα. Εν συνεχεία, έπρεπε να οργανώσουμε τη δουλειά αυτή με τα κράτη-μέλη, γιατί οι εκλογές είναι πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών. Ε, στο εκλογικό πακέτο, λοιπόν, εντοπίσαμε μία σειρά από μέτρα. Ένα σημαντικό μέτρο είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο έγκαιρη προειδοποίηση, δηλαδή με σημεία επαφή στα κράτη-μέλη που θα ενημερώνουν ο ένας τον άλλον, το ένα ε, σημείο επαφής θα ενημερώνει του ομοτήμού του α πούμε, ε, για τους ε, κινδύνους που αφορούν όλη την Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν αυτό το δίκτυο, υπάρχει αυτό το σύστημα και λειτουργεί πλήρω τώρα. Το άλλο σύστημα συνεργασίας που δημιουργήσαμε στα πλαίσια τη Οδηγία για την Κυβερνοασφάλεια είναι μια ομάδα συνεργασία για την κυβερνοασφάλεια ενώπιση των εκλογών. Αυτή τη εβδομάδα θα γίνει μια άσκηση η οποία με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δοκιμάσουμε την κυβερνοασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας ε, που αφορούν τις εκλογές. Και δουλεύουμε με τους ε, εμπειρογνωμόνους των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπολείπων θεσμικών οργάνων για να εξασφαλίσουμε την κυβερνοασφάλεια κατά εκλογές. Ένας άλλος σημαντικός τομέας εργασίας είναι ε, να συνεργαστούμε με οργανώσεις που ελέγχουν τα δεδομένα, τα στοιχεία. Είναι περίπλοκο αυτό, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε οργανώσεις τις οποίες ε, σπονσοράρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν είναι στοιχείο ανεξαρτησίας αυτό. Θέλουμε να είναι πραγματικά ανεξάρτητες αυτές οι οργανώσεις, ε, αξιόπιστες και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι ότι δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα όπου μέσω της οποίας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις στατιστικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, την βάση δεδομένων της Eurostat, το καταθετήριο ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, με τις δημοσιεύσεις και το δικό μας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Έχουμε πάνω από 80 τέτοιου οργανισμούς που ελέγχουν τα δεδομένα και που συμμετέχουν στην πλατφόρμα και είναι στο περισκόπιό μας και θα πάμε στην επόμενη φάση θα χρησιμοποιήσουμε χρηματοδότηση από το Europe Connecting Facility, από το Μηχανισμό Συνδέοντα την Ευρώπη, για να οργανώσουμε αυτό το δίκτυο ακόμα πιο διαρθρωμένα. Όχι χρηματοδοτώντα απευθεία τι οργανώσει αυτέ ελέγχου των δεδομένων, αλλά εξασφαλίζοντα εξασφαλίζοντάς τους όλα τα εργαλεία, ούτως ώστε να δουλέψουν καλύτερα και να συνεργαστούν μεταξύ τους καλύτερα. Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα στο οποίο προβαίνουμε. Ε, μίλησα ήδη για τη γνώση των ε, μέσων ενημέρωσης ε, και τα όσα προβλέπει η οδηγία για τα οπτικοακουστικά. Υπάρχει αυτό το νέο στοιχείο του literacy της ε, οδηγίας και που είναι η δημιουργία στην Ευρώπη ε, ασφάλειας δικαίου ότι θα υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές ανεξάρτητες για τα μέσα ενημέρωσης. Ό,τι εφαρμογή και να κάνει κανείς, θα πρέπει να έχουμε την εγγύηση ότι αυτές οι οργανώσεις είναι ανεξάρτητες από τις κυβερνήσεις. Γιατί αυτό το θέμα ή και άλλα θέματα μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν και να χειραγωγήσουν η εκτελεστική εξουσία, οι κυβερνήσεις δηλαδή. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. θα πρέπει η ομάδα των εξάρτητων ε, ρυθμιστικών αρχών που έχουν και ε, νομικό καθεστώς υπό την οδηγία για τα οπτικοακουστικά να μας, ε, να μας υποστηρίζουν αναλύοντας τα αποτελέσματα του κώδικα δεοντολογίας και εκεί ε, συνεργαζόμαστε με τους ανεξάρτητους αυτούς ρυθμιστικούς φορείς, το έργα. Ε, ας πούμε στη Γαλλία και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες ε, δια νόμου ελέγχουν ε, την αξιοπιστία των επικοινωνιών κατά τις εκλογές. Έχουν δηλαδή ε, αρμοδιότητες δια νόμου. Όσο προβάλλουμε στο μέλλον. Θέλουμε να έχουμε εγγυήσεις ότι υπάρχει πραγματικά ανεξάρτητη αξιολόγηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα περνάω σε ένα άλλο θέμα. Μίλησα ήδη για το literacy, για το, τη γνώση των μέσων. Ε, ένα άλλο θέμα είναι οι ρητορίες μίσους, η καταπολέμηση του ρατσισμού στο διαδίκτυο και άλλα προβλήματα που αποτελούν προσβολή για την κοινωνία. Αυτό είναι τμήμα της νέας του εργαλειοθήκης ε, για τις οπτικοακουστικές ε, υπηρεσίες. Και αυτό γίνεται με ένα τρόπο ούτως ώστε την πρώτη ευθύνα να την έχει η πλατφόρμα, αλλά η συνεχεία μπαίνουν και οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές και υπάρχει και ένας μηχανισμός αναφοράς παραπώνων. Ε, όταν βλέπουμε τους κανόνες το πρώτο που θα πρέπει να έχω στο μυαλό μας είναι ότι υπάρχει μια ολοκένουργια οδηγία για τα οπτικοακουστικά που θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτή η οδηγία ήδη προβλέπει ε, πολύ σημαντικά νέα εργαλεία για το σεβασμό των βασικών αρχών ε, για τα ΜΜΕ στην Ευρώπη. Βραχυπρόθεσμα λοιπόν, κάναμε μια πολύ σημαντική δουλειά ε, που έχει αναγνωριστεί από το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά εν συνεχεία γίνεται μια πολύ πιο περίπλοκη συζήτηση για το τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Φυσικά εδώ μπαίνει και το νέο κοινοβούλιο, στη νέα του σύνθεση δηλαδή, ε, και ο νέος θεσμικός κύκλος που θα παίξει το ρόλο του. Αυτά που κάναμε εμείς ήταν η αφετηρία. Το βασικό ερώτημα θα, ήταν, θα είναι τώρα αν αυτέ οι μορφέ αυτορύθμιση είναι αποδοτικέ αν λειτουργούν ή όχι. Και φυσικά, με μεγάλη χαρά θα συνεισφέρουμε στην νέα αυτή συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει, εάν κάτι πρέπει να γίνει δια νόμου, μέσω νομοθεσία, λαμβάνοντα υπόψη όλα τα στοιχεία ε, τα οποία έχουμε μέχρι στιγμή στη διάθεσή μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βιόλα. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά μας ε, σημεία στις συζητήσεις που είχαμε για αυτή την οδηγία. Είχαμε την βούληση να υπάρχουν συστήματα αυτορύθμισης και να τα ενισχύσουμε, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα εγκατασταθούν και αν πραγματικά επιφέρουν τις επιτυχίε τις οποίες επιθυμούμε και ε, στο εγγύς ε, μέλλον να δούμε αν ο κώδικας ο οποίος έχουμε αναπτύξει είναι έτσι τόσο ώστε να πούμε ότι πραγματικά μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις ψευδείς ειδήσει, την παραπληροφόρηση, να τις περιορίσουμε και βλέπω τώρα ότι έχει ζητήσει ε, ο κύριος Τούρλ τον λόγο. Η κυρία Τούρλ. Ευχαριστώ πολύ πιστεύω ότι είναι επίγον να συζητήσουμε το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων και ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ψευδείς ειδήσει υπήρχαν ανέκαθεν. Όμως ε, η διανομή τους μέσω του ίντερνετ ε, έχει, γίνεται πλέον σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Μετά την ορκομοσία του, ο Ντόναλτ Τραμπ ε, είχε πει όταν δεν ήταν ικανοποιημένο από το κοινό που είχε βγει στου ε, δρόμου, ε, είχε πει αυτά είναι εναλλακτικά δεδομένα, alternative facts. Έτσι λοιπόν μιλάμε για αυτά τα εναλλακτικά δεδομένα. Δεν το πιστεύω αυτό. Υπάρχουν, υπάρχει πραγματικότητα και η ε, σωστή δημοσιογραφία μιλά για την πραγματικότητα φυσικά και υπάρχουν διαφορετικές ε, απόψεις, όμως θα πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην γνώμη και στην δημοσιογραφία. Όμως αυτό πλέον έχει ε, μπερδευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των δύο. Ένα παράδειγμα με την περίπτωση του Christchurch. Γνωρίζετε ότι αναμεταδόθηκε ζωντανά και ουσιαστικά προωθούσε την τρομοκρατία. Στην συνέχεια άσκησα κριτική για αυτό στο Twitter αλλά και στην ε, γερμανική τηλεόραση και ισχυρίστηκα ότι μετά το Christchurch η εντύπωσή μου είναι ότι προφανώς ε, και χρειαζόμαστε ορθούς κανόνες για τα μέσα μαζικής ε, δικτύωσης. Δεν το συνδέσα, συνέδεσα με το άρθρο 13 τότε και στη συνέχεια στο Twitter δέχθηκα επιθέσεις ότι χρησιμοποιούσα νεκρούς για να προωθήσω το άρθρο 13. Δεν ήταν αυτό όμως το επιχείρημά μου. Το ε, ένα αφορούσε τη μεταρρύθμιση για το copyright και ε, το άλλο ήταν εντελώ διαφορετικά τα θέματα. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι μετά το Christchurch θα πρέπει να λάβουμε δράση και τώρα καλούνται οι πολιτικοί να θεσπίσουν ορθούς κανόνες και στη συνέχεια υπήρχαν νέοι στο ίντερνετ οι οποίοι είπαν όμως η τηλεόραση έκανε ακριβώς το ίδιο ανέφεραν τα όσα συνέβησαν εκεί και δεν κατανοούμε την διαφορά ότι αν το προωθείς κάτι ζωντανά ως τρομοκρατία και όταν το αναφέρει τηλεόραση είναι δύο διαφορετικά πράγματα και οι πολίτες πολύ συχνά δεν αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο. Θεωρώ ότι γενικά θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ψευδείς ειδήσει με μη ψευδείς ειδήσει. Ε, υπάρχει αυτή η ποικιλομορφία ε, πληροφοριών και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τι είναι ψευδές και τι όχι. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίε. Ε, και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε τις ψευδείς ειδήσει. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ζητήσουμε από τι εταιρείε και από τα μέσα κοινωνική Για πολλά χρόνια ε, λέγανε το YouTube για παράδειγμα ότι απλά μεταφέρει ε, βίντεο, ειδήσει, όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι επηρεάζεται με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Χέλγα. Είναι η τελευταία μας συνεδρίαση, όμως παρόλα αυτά θα πρέπει να κοιτάμε και το ρολόι, να μην ξεφύγουμε. Οπότε θα πρέπει να περιοριστούμε όλοι στα 2-3 λεπτάκια και θα τα καταφέρουμε. Κυρία Κώστα. Ευχαριστώ το Γενική, Γενικό Διευθυντή για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε η Γενική σας Διεύθυνση με τις 17 πρωτοβουλίες ε, που μας έφεραν σε ένα καλό σημείο. Νομίζω ότι όλο το σύστημα του ευρωπαϊκού αυτού συναγερισμού είναι πολύ σημαντικό. Τα κοινωνικά μέσα ε, διαδίδουν ειδήσει ε, όλο και περισσότερο με εκθετικό χαρακτήρα και εμείς τρέχουμε από πίσω, προχωράμε βέβαια. Ε, μιλάμε τώρα για μέσα κοινωνική δικτύωσης όπου ε, εκτός από το hate speech, εκτός από τις ρητορίες μίσους κτλ. έχουμε και προσωπικές επιθέσεις που οδήγησαν ας πούμε σε αυτοκτονίες. Έτσι, ε, γιατί κάνουν ε, αξιολογικές κρίσεις και λανθασμένα πράγματα λένε για τα άτομα. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε μεγάλη σχέση με την επιστημονική κοινότητα για να έχουμε σωστές πληροφορίες. σας. Είναι σημαντικό ο κώδικας δικοντολογίας, ο μηχανισμός ε, έγκαιρης απάντησης τα focal point, τα, σημεία, τα εστιακά σημεία, τα σημεία σύνδεση που είναι στα κράτη-μέλη, όλο αυτό το σύστημα αρχιτεκτονική για να έχουμε ένα συντονισμό ε, παρεμβάσεων και απαντήσεων. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, εγώ δεν πιστεύω πολύ στα συστήματα αυτορύθμισης όταν παίζουν, μπαίνουν εδώ ουσιαστικές αξίες της ένωση Θα πρέπει να τσεκάρουμε αν λειτουργούν. Στην πρώτη έκθεση που έγινε τον Ιανουάριο στους τρεις επιτρόπους από τις πλατφόρμες. Υπήρχαν τρομερά ελλείμματα, καθυστερήσεις και δεν υπήρχε πραγματική βούληση να απαντήσουν οι πλατφόρμες σε όλες τις ερωτήσεις των τριών επιτρόπων. Δεν θα πρέπει να ε, μείνουμε μόνο στα, στην αυτορύθμιση, θα πρέπει να υπάρχει, υπάρξει και ρύθμιση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με τις αξίες και τα δικαιώματα. Επίσης, ε, έχουμε Μία δράση σε τρεις πυλώνες. Σωστό. Γίνεται κάτι για τις ε, εκστρατείες παραπληροφόρησης. Η, γιατί η Wikipedia κάνει τέτοια εκστρατεία παραπληροφόρησης. Ε, έχει μία στάση που διαμορφώνει την άποψη των ε, χρηστών για μία οδηγία του Κοινοβουλίου ε, και την ε, διαμόρφωσε με βάση fake news. Ε, δημιουργούνται αυτά τα fake news για οικονομικούς λόγους και διαμορφώνουν τη δημόσια συζήτηση. Ε, όμως προωθούνται τα fake news με έναν τρόπο πάρα πολύ προχωρημένο και επηρεάζουν και τις απόψεις μας και την υγεία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε. Σημερίζομαι την άποψη ότι έχουμε καθυστερήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε μια πολύ σημαντική ψηφοφορία σχετικά με το copyright και θα ήθελα να μου πείτε τι γνωρίζει η Επιτροπή σχετικά με τις εξωτερικές ε, δραστηριότητες, ε, σχετικά με τις προσπάθειες που γίνονται ε, για την επιρροή των ευρωβουλευτών ή το λόμπι που εκτελήθηκε ήταν ιδιαίτερα έντονο. Εμείς καθυστερήσαμε όσον αφορά τα αντιμέτρα και το κέρδος της γνώσης ε, λοιπόν. Οπότε το ερώτημά μου είναι τι ακριβώς γνωρίζουμε σχετικά με τα αίτια των ψευδών ειδήσεων, τους ε, συγγραφείς τους, ε, αλλά και τις συνέπειες που έχουν αυτές οι ειδήσει. Διότι έτσι θα μπορούμε στη συνέχεια να αξιολογήσουμε τα μεμονωμένα μέτρα τα οποία λαμβάνονται Κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις ε, σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ακούσαμε ότι δαπανώνται εκατομμύρια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και όσοι διανέμουν ε, ψευδείς ειδήσεις από την άλλη δαπανούν δισεκατομμύρια. Οπότε γίνεται το ερώτημα ποιος ακριβώς είναι αυτός ο παραγωγός των ε, ψευδών ειδήσεων, πόσο μεγάλο είναι το εύρος τους, ποιος ακριβώς βρίσκεται από πίσω, ποιες οργανώσεις ε, υπάρχουν και κρύβονται από πίσω και κατά πόσο οι ευρωβουλευτές μπορούν ε, να ελπίζουν ότι θα υπάρχει προστασία από τις δραστηριότητες των λόμπι που είναι ιδιαίτερα επιθετικές ε, και ασκούν μεγάλη πίεση. Ευχαριστώ ε, πολύ. Ο κύριος Ποσταμίτη. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Βιόλα, όπως και οι συναδελφοί μου, για την ε, παρουσίασή σας. Αναφερθήκατε σε τρία είδη ψευδών ειδήσεων όσον αφορά την αποστεθροποίηση της δημοκρατίας, αυτοί οι οποίοι θέλουν να διασπείρουν τον πανικό ε, και ε, η χειραγώγηση των γνώμεων. Η κατάσταση είναι πολύπλοκη διότι οι διάφοροι τομείς αυτοί μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται κάτι το οποίο είναι μια άποψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία μας και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η μάχη μας κατά των ψευδών ειδήσεων θα πρέπει να ενισχυθεί διότι η ίδια η δημοκρατία μας βασίζεται στο ότι λαμβάνουμε ενημερωμένες αποφάσεις και όταν οι αποφάσεις αυτές είναι ε, λανθασμένα ενημερωμένες τότε και όλη η διαδικασία λήψης απόφασης ε, ε κινδυνεύει. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν συμφωνώ μαζί σας πως όταν μιλάμε για δομές εντός των κρατών μελών που θα πρέπει να μας προστατεύουν, οι δομές αυτές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες, διότι το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι δομές οι οποίες βασίζονται στην εκτελεστική εξουσία, όπου οι κυβερνήσεις αποφασίζουν τι είναι αληθές και τι όχι. Οι κυβερνήσεις άλλωστε δεν είναι και ε, πάντοτε αθώες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης ε, για πρωτοβουλίες σχετικά με την προώθηση των ε, μέσων, ε, προσπάθειες έχω ακούσει ότι έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες από ανεξάρτητους fact-checkers και η συζήτηση σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις θα πρέπει επίσης κατά τη γνώμη μου να, να συνδεθεί και με τη συζήτηση για τη χρήση προσωπικών δεδομένων διότι στο, ο Ντέιβις στο έργο του Post-Truth έχει μιλήσει ότι όλοι έχουμε την προκατάληψη της επιβεβαίωσης και υπάρχουν ε, ε υπάρχουν προφίλ τα οποία γνωρίζουν τι προκαταλήψεις έχουμε όπως ε, ε, συνέβη με την Cambridge Analytica και αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο σε μαζικό επίπεδο αλλά και σε μικροεπίπεδο και θα ήθελα να αναφέρω ότι προσφάτως είχα συναντήσει με Google και Facebook ε, σχετικά με το ζήτημα της αυτορύθμισης, όμως ακόμα διαρκεί πολύ και γι' αυτό το λόγο θα χρειαστούμε πιο γρήγορα μέτρα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σκόρντοβα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι έχουν καλύψει τα πιο σημαντικά σημεία. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις ψευδείς ειδήσει. Σίγουρα πρέπει να στηρίξουμε την κριτική σκέψη, τη γνώση και το γραμματισμό όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών και η κριτική σκέψη είναι κάτι το καθοριστικό. Δεν είναι εύκολο, το ξέρουμε όλοι. Πώς μπορεί κάποιος να εντοπίσει τις ψευδείς ε, ειδήσει. Και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Ας κοιτάξουμε τα διάφορα θέματα τα οποία στοχεύουν αυτές οι ψευδείς ειδήσει. Είναι κυρίως θέματα που δεν γνωρίζουν καλά οι πολίτες. Είτε παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί δεν έχουν έρθει να δουν πώς λειτουργούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν έρθει να δουν πώς δουλεύουμε. Το καλύτερο λοιπόν είναι να υπάρξει επαλήθευση, να γνωρίζει κανείς την πραγματικότητα, πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόληψη λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντική για να υπάρξει εμπιστοσύνη στη λειτουργία μας. Πολύ σύντομα η Τζούλι Θα είμαι πολύ σύντομη. Καταρχήν η χώρα μου είναι ένα από τα θύματα αυτών των ψευδών ειδήσεων και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος μας έδειξε ότι πολύ αργά σήμερα αντιλαμβανόμαστε, αντιλαμβάνονται πολλοί στη χώρα μου ότι υπήρξαν θύματα παραφληροφόρησης. Συμφωνώ με συναδέλφους που είπαν ότι χρειάζεται πολύ καλύτερη ε, χρήση αυτών των δεδομένων και ότι στην Ευρώπη, αλλά μιλώ κυρίως για τη δική μου χώρα, δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Οι πολίτες μας δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, δεν ξέρουν ότι δικαιούνται σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση. Και πέρα από τη γνώση του ψηφιακού κόσμου, από τη γνώση των τεχνολογιών και του διαδικτύου, νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί στους νέους τουλάχιστον μία πιο έντονη κριτική σκέψη. Να τους κινήσουμε την περιέργεια και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερο από σωστές πηγές. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι ακριβώς οι ψευδείς ειδήσει, τι είναι η παραπληροφόρηση, τι είναι οι λόγοι μίσους, η παρότρινση σε ρατσισμό, ξενοφοβία και η παραπληροφόρηση δεν είναι κάτι που τιμωρείται από τον νόμο, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς πού σταματάει η παραπληροφόρηση, πού αρχίζουν οι σκόπιμα ψευδές ε, ειδήσει και πού ε, υπάρχουν οι αξιόπινες πράξεις όπως ε, οι λόγοι μίσους και η παρότρινση σε φανατισμό και ρατσισμό. Σίγουρα θα πρέπει να στηρίξουμε την ποιοτική δημοσιογραφία, η κατάρτιση των δημοσιογράφων οι δημοσιογράφοι δεν θα πρέπει να εξετάζονται και να καλούνται να έχουν μόνο δεξιότητες όσον αφορά τη δημοσιογραφία αυτή καθεαυτή, αλλά να μπορούν να επαληθεύσουν και να εντοπίσουν τις πηγές ε, όταν βασίζονται σε κάποιες πληροφορίες για να γράψουν κάποιο άρθρο, για να διαδώσουν κάποιες ειδήσει. Μιλήσατε για 80 ανεξάρτητους φορείς και οργανώσεις. Δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπίσει κανείς ε, τις εσφαλμένες ειδήσει, αλλά πρέπει να βασιζόμαστε σε πραγματικά περιστατικά και βεβαίως δεν θα πρέπει να στηρίζουμε οικονομικά κάποιους οργανισμούς που ξέρουμε ότι δεν είναι ανεξάρτητοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τον εντοπισμό αυτών των ανεξάρτητων φορέων. Θα πρέπει να συνεχίσει να τους στηρίζει γιατί παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία μας. Κύριε Βιόλα, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Όλα τα μέλη που πήραν το λόγο ε, έχουν συνεισφέρει με πολύ σημαντικό τρόπο στη συζήτηση αυτή. Βεβαίως δεν μπορώ να σχολιάσω όλα αυτά που άκουσα. Θα προσπαθήσω να εντοπίσω σε κάτι που νομίζω ότι άκουσα σχεδόν από όλους τους ε, παρεμβαίνοντες. Είναι αλήθεια και εδώ συμφωνούν και οι δημοσιογράφοι και οι δικαστές και οι επιστήμονες και οι κοινωνιολόγοι αυτό που είναι, αν θέλετε, αλήθεια, επιστημονική αλήθεια, διαπιστώνουμε ότι στους δημοσιογράφους πολλές φορές, παρόλο που οι πηγές τους είναι πηγές συνήθως που επαληθεύονται, δεν μεταφράζονται με τον ίδιο τρόπο. Η πραγματικότητα, η πραγματικότητα είναι αυτή και γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ποιοτική δημοσιογραφία. Αν κοιτάξει κανείς τους πιο δυνατούς φορείς και εταιρείε στον κόσμο, διαπιστώνουμε ότι η ευθύνη δεν επικρατεί στις επιχειρήσεις αυτές. Βεβαίως πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανεκτικοί όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μία εταιρεία που μόλις ιδρύθηκε, μια startup. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε εξίσου ανεκτικοί και να δείχνουμε ανοχή όταν υπάρχει παραβίαση των κανόνων από μέρους των μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων. Αυτό που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εξαιρετικά σημαντικό, η οδηγία για την μεταρρύθμιση των οπτικοακουστικών μέσων. Η πρόοδος αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και παραδείγματο χάρη να κοιτάξει κανείς αυτό που συνέβη στο Christchurch. Σαφώς ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά, αλλά εδώ θα πρέπει να εντοπιστούν οι ρυθμιστικές αρχές, ποιος είναι ο ρόλος τους και τι ε, κενά υπάρχουν. Οι κανόνες λοιπόν υπάρχουν στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει πολύ σημαντικούς κανόνες. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Επίσης, το θέμα των πλατφόρμων. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει οθετήσει πολύ σημαντικούς κανόνες το θέμα των συμφωνιών που έχουν οι πλατφόρμες αυτές με επιχειρήσεις και φορείς. Θα πρέπει να επικρατεί διαφάνεια, να είναι γνωστές οι συμφωνίες αυτές, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κατονίσουμε καλύτερα πώς επεξεργάζονται τις πληροφορίες. Οι σχέσεις λοιπόν μεταξύ πλατφόρμας και επιχειρήσεων είναι κάτι που θα πρέπει να το επεξεργαστούμε περισσότερο. Επίσης, το θέμα της ανεξάρτητης επαλήθευσης των γεγονότων, των περιστατικών και των δεδομένων. Υπάρχουν ανεξάρτητοι φορείς που ελέγχουν τα δεδομένα. Εμείς δεν στηρίζουμε αυτούς τους φορείς. Δεν είναι ο ρόλος μας. Αλλά έχουμε δημιουργήσει το πλαίσιο αυτό μέσα στο οποίο μπορούν να λειτουργήσουν ανενόχλητοι. Και βεβαίως εδώ υπάρχει και η βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Βεβαίως λοιπόν στηρίζουμε την ποιοτική δημοσιογραφία στο νέο πρόγραμμα για την Δημιουργική Ευρώπη. Δεν υπάρχει αναφορά στην ποιοτική δημοσιογραφία. Υπάρχει όμως ένα ποσό 80 εκατομμυρίων ευρώ που θα στηρίξει τον τομέα αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βιόλα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα το πρωί που μας ενημερώσατε για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι πεπισμένη ότι και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ασχολείται, θα πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα αυτό, διότι δεν πιστεύω ότι σε έξι μήνες τα πράγματα θα έχουν βελτιωθεί. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσία σας, σα ευχαριστώ πολύ για τι προσπάθειές σα για την παρουσίασή σα. και ελπίζω πραγματικά όλα αυτά θα υλοποιηθούν. Ελπίζω ο κώδικας ε, δεοντολογίας, ο κώδικας ορθής πρακτικής θα εφαρμοστεί και ελπίζουμε πραγματικά να έχουμε αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να στηρίζουμε την ποιοτική δημοσιογραφία. Πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε αυτό. Επαναλαμβάνω ότι από τον υπιαγωγείο και όλα θα πρέπει να ξεκινάει αυτή η συνείδηση, η κριτική σκέψη και νομίζω ότι όλο αυτό το φάσμα μέτρων και οι διάφορες μέθοδοι εργασίας που έχουν υιοθετηθεί αλλά και παραπάνω ρύθμιση θα μας βοηθήσουν να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια και βεβαίως μπορείτε να παραμείνετε μαζί μας. Δεν ξέρω αν σας ενημέρωσαν ότι έχουμε οργανώσει ένα μικρό κοκτέιλ και είστε ευπρόσδεκτος. Σας ευχαριστώ πολύ. So, liebe Kolleginnen Αγαπητοί Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα αναπροσαρμοστούμε λιγάκι εδώ. Thank Petra. Hi. So, jetzt bin ich hier im falschen, falschen Text gelandet. Ich freue mich sehr zum nächsten Tagesordnung. Χαίρομαι ιδιαίτερω για το επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, το οποίο αφορά τη συζήτηση σχετικά με την κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους ε, Πολιτιστική ε, κληρονομιάς. Ε, έχουμε την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης ε, ΕΑΚ μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Η χρονιά αυτή ήταν ε, μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της, του Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να πούμε ότι και όσον αφορά την εφαρμογή του ήταν μια μεγάλη επιτυχία το οποίο φαίνεται από τις αναρρύθμιτες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς καθώς επίσης και το μεγάλο αριθμό των πολιτών που συμμετείχαν. Θα επιθυμούσα η ευρωπαϊκή χρονιά να ήταν λιγάκι πιο ευρωπαϊκή διότι πολλές δραστηριότητες ε, εν μέρη επικεντρώθηκαν ε, στο εθνικό κομμάτι. Παρόλα αυτά όμως ε, πιστεύω ότι ήταν μια επιτυχία διότι ο πολιτισμός ήρθε στο επίκεντρο της συζήτησης και κατά την άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το momentum που δημιουργήθηκε πέρσι διότι θα ήταν κρίμα εάν αυτή η βασική θέση που έλαβε στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πολιτισμικό στοιχείο, ε, εάν χαθεί αυτή η ευκαιρία. Και θα ήθελα να πω ότι ήμασταν λιγάκι απογοητευμένοι όταν είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά την ανακοίνωση σχετικά με το πολιτιστικό έτος δεν έκανε ε, μία ανακοίνωση ε, και εν τέλει περιορίστηκε μονάχα σε ένα ε, έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο μου δίνει την αίσθηση ότι η βιωσιμότητα του πολιτιστικού έτους βρίσκεται μάλλον προς το τέλος της στο τέλος του θεματολογίου της Επιτροπής και γι' αυτόν τον λόγο ε, χαίρομαι που τώρα θα κάνουμε μία συζήτηση με την ελπίδα ότι το έτος αυτό ίσως να ενισχυθεί κάπως ε, και ε, να έχουμε διευκρινήσεις και εξηγήσεις πάνω στις ανησυχίες μας και ότι η Επιτροπή θα θέσει φιλόδοξους στόχους με τους οποίους θα μπορέσει να ασχοληθεί το επόμενο Κοινοβούλιο. Κυρία Χριστοφίδου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ, θέλω να σας καθησυχάσω καταρχάς. Αισθάνομαι ότι αν κοιτάξετε την ομάδα στην ε, Γενική Διεθνή Άκτα που ασχολήθηκε με αυτό το ε, έτος, θα δείτε ότι ασχοληθήκαμε με πάθος και με ενθουσιασμό και αυτό θα σας καθησυχάσει για το κατά πόσο μας ενδιαφέρει και το πόσο βιώσιμο είναι αυτό το project. Εάν ε, έχει να κάνει με εμά, προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι, θα, τι συνέχεια θα δοθεί στο έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Εγώ έφυγα από την πατρίδα μου πολύ μικρή και η σχέση μου με την Κύπρο, την πατρίδα μου, ε, αισθάνομαι ότι εξαρτάται από την διασφάλιση της ε, κληρονομιάς μας. Από τα στοιχεία, ε, τα υλικά στοιχεία, ας πούμε, αυτής της κληρονομιάς που κουβαλάμε μαζί μας. Εγώ στα 12 μου έφυγα ε, το 1974 από την ε, πατρίδα μου και παρότι παρέμεινα στον ίδιο κόσμο Εβραίος πως ε, δεν είχα την ιδιαίτερη πατρίδα μου, δεν είχα το ψωμάδικο, ε, το θέατρο, ε, τις γιορτές το Πάσχα, ακόμα και τις ίδιες οικογενειακές φωτογραφίες. Θέλουμε να διατηρήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά και το θέλουν όλοι. Και αυτό το καταλαβαίνω, όχι μόνο ως Γενική Διευθύντρια της Κομισιόν, αλλά και ως άτομο, εγώ, η Θέμης. Ε, είναι έκφραση της συλλογική μας μνήμης, που θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή αυτή η πολιτιστική κληρονομιά. Ε, με, ως μέλος της πόλης μας, της περιοχής μας, ε, της χώρας μας, της Ευρώπης μας. Το να χρησιμοποιήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά μας βοηθάει να καταλάβουμε τον εαυτό μας καλύτερα και τους άλλους καλύτερα. Ε, βλέπουμε, αγγίζουμε, γευόμαστε τους άλλους ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικές παραδόσεις και άλλες χώρες και μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς αυτές οι διαφορές είναι πολύτιμες, γιατί υπάρχει ομορφιά ε, εκεί ε, και ιδιοφία. Αυτή η κοινή κατανόηση ε, μιας κοινωνίας που γιορτάζει τον πολιτισμό της άλλης κοινωνίας χωρίς φόβο για τη διατήρηση της δικής της ε, κληρονομιάς είναι η κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το ευρωπαϊκό έτος ήταν μια αναμφισβήτητη επιτυχία. Πάνω από 18.000 εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν το 18 σε όλη την Ευρώπη, ε, όπου συμμετείχαν πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωπα. 30 εκατομμύρια συμμετείχαν στην δική έκδοση της, των, της ημερίδας ε, Ευρωπαϊκής ε, Πολιτικής Κληρονομιάς. Ε, είχαμε διάφορες, 14.000 έργα, project, εκδηλώσεις. Αυτό είναι το συλλογικό μας επίτευγμα. Χωρίς τη στήριξη και την επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα υπήρχε τέτοιο ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς καθόλου, το ξέρουμε και σας είμαστε ευγνώμονες. Μην ξεχνάτε εσείς τα μέλη αυτής της Επιτροπής και ειδικά εσείς κυρία Πρόεδρε, κυρία Κώστα, Διακόνου, κυρία Σόιντοβα, ήσασταν και είσαστε ε, σύμμαχοί μας ενεργό ρόλο στις αστριότητες του 18 και οργανώσατε και αξιομνημόνευτες εκδηλώσεις όπως ας πούμε ε, τον Ιούνιο στο ημικύκλιο ε, την ε, εκδήλωση υψηλού επίπεδου και τη συνάντηση τον Νοέμβριο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Με αυτόν τον τρόπο προωθήσαμε τους στόχους της πολιτικής μας. η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μπήκε ψηλά στην πολιτική ατζέντα, στο πολιτικό θεματολόγιο της Ευρώπης. επηρεάσαμε επίσης ε, το πώς βλέπουν οι φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς ε, την ιστορία αυτή. Ε, κάθε project είχε τις δικές του αξίες, όχι μόνο γιατί γιορτάζει την τέχνη της Ευρώπης σε όλη την ποικιλομορφία της, αλλά και γιατί φέρνει κοντά τους ανθρώπους που εκφράζουν τους πολίτες της Ευρώπης στο παρελθόν, στο παρόν και, στο... και για πολλά χρόνια στο μέλλον. Ε, η φιλοδοξία μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι η ατμομηχανή για την ε, διασφάλιση και τη διατήρηση της δικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς αυτή. Η φιλοδοξία είναι η βάση του, της χρονιάς του 18 και του σχεδίου ε, follow-up 15 υπηρεσίες της Κομισιόν συνεργασία με τα κράτη-μέλη και με ο, φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς ε, προωθούν 65 ε, δράσεις ε, μέσα στο 2019 και το 2020. Το πλαίσιο δράσης για τη συμμετοχή όλων, όπου διονύζουμε την παράδοση για την έμφαση στην ποικιλομορφία. Εξάλλου αυτό μας φέρνει κοντά και έχει σημασία για όλους μας. Επομένως, ο καθένας, όσο διαφορετικός και αν είναι, θα πρέπει να συμμετέχει. Υπ' αυτή την έννοια συνεχίζουμε να προωθούμε τις ε, συμμετοχικές πρωτοβουλίες όπως ε, οι μερίδες ε, ευρωπαϊκής κληρονομιάς καθώς και η όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση, ψηφιακή πρόσβαση μέσω της Ευρωπαϊάνα. Όλοι οι φορείς ε, επίσης εμπλέκονται. μια συνεργασία ε, multi-stakeholder με πολλούς φορείς δηλαδή ήταν κλειδί για την επιτυχία της χρονιάς. Υπάρχει και ένα φόρουμ, μια ομάδα εμπειρογνωμών της Κομισιόν για να εφαρμόσουμε το πλαίσιο αυτό για δράση της Κομισιόν. Ε, οι εκπρόσωποι εκεί των κρατών μελών, ε, ο πρόεδρος λέει να μιλάει λίγο πιο αργά η ομιλήτρια, αλλά εγώ είμαι αγχωμένη, λέει, γιατί φοβάμαι θα μου κόψετε το λόγο. Ε, η πέτρα είναι πολύ σκληρή και με αγχώνει. Εκεί ακριβώς οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών θα δώσουν τη δική του συνεισφορά. Τρίτον, η κληρονομιά δεν είναι, διαφορετική, δεν είναι ανεξάρτητη από την καθημερινότητά μας. Η κληρονομιά μας αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε προγράμματα και πολιτικές, αλλά θα πρέπει να συνεισφέρει ενεργά σε έξυπνες λύσεις όταν είναι χρήσιμα σε αυτές. Φερρυπίν, η κληρονομιά έχει σημαντικό ρόλο στην διεθνή συνεργασία στο να βοηθήσει την Ευρώπη να δημιουργήσει ε, σταθερούς δεσμούς με άλλα μέρη του κόσμου. Ένας άλλος σημαντικός τομέας είναι η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Η αστική ατζέντα, το αστικό θεματολόγιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίνει σημαντική θέση στον πολιτισμό και στην πολιτιστική κληρονομιά με ένα νέο εταίρο ε, που, με μια εταιρική σχέση που ξεκίνησε στο Βερολίνο τέλη Φεβρουαρίου. Εκεί οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, ε, διάφορες εταιρείες από τις πόλεις και τους δήμους ε, συνέρχονται και η εταιρική σχέση θα ετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης για βασικά θέματα που σχεδέονται με τον πολιτισμό και την ε, κληρονομιά στις ευρωπαϊκές πόλεις για βελτίωση της νομοθεσίας, της χρηματοδότησης και τον επιμερισμό της γνώσης. Τέταρτον, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την κληρονομιά που κινδυνεύει, να προωθήσουμε τη βιωσιμότητά του και να υποστηρίξουμε τους επαγγελματίες του κλάδου. Ένα άλλο σημαντικό καθήκον είναι να αντιμετωπίσουμε το λαθρεμπόριο ε, πολιτιστικών αγαθών και να εξασφαλίσουμε αρχές ποιοτικέ για χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στοιχείων του πολιτισμού. Ε, καλωσορίζω τα θετικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου για τον κανονισμό για την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον περασμένο μήνα, δηλαδή χώρα αυτή η, η ψηφοφορία. Πέντε, θα κινητοποιούμε τη γνώση και την έρευνα για τεχνική και κοινωνική καινοτομία για την κληρονομιά με την υποστήριξη του ορίζοντα 2020 και το νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία. Το 2018, ο ορίζοντας 2018 ε, επένδυσε 66 εκατομμύρια για έρευνα σε πολιτιστική κληρονομιά που είναι ένα πολλαπλάσιο από αυτό που, που είχαμε στο Creative Europe. Ε, ο ορίζοντας Ευρώπη θα πρέπει να κρατήσει, το Horizon Europe θα πρέπει να κρατήσει το ίδιο επίπεδο φιλοδοξία τουλάχιστον. Θέλουμε αυτό το πλαίσιο πολιτιστική να υποστηριχθεί από καλή χρηματοδότηση και αυτό είναι στοιχείο κλειδί. Στο, στην ε, μελλοντική πρόταση της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό προβλέπουν ένα συνολικό προϋπολογισμό 1,85 δις ευρώ. Όμως η στήριξη για την πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να είναι ακόμα ευρύτερη. Ε, οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό συνεχίζονται και βασιζόμαστε ακριβώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας, ούτως ώστε να υποστήριξει το επιχείρημα ότι έχει σημασία ε, να στηρίξουμε τον πολιτισμό πέρα από το πρόγραμμα της Δημιουργικής Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για την, τον ενθουσιώδη, την ενθουσιώδη συμμετοχή σας, για αυτή την πολύ εντυπωσιακή χρονιά. Ε, το είπα βέβαια όταν είναι θαυμάσια και μοναδική επιτυχία. Θέλω να το ξαναπώ. Ε, κανονικά ήταν καταλήτης για να, είναι, ε, για να προωθήσει τις τοπικές, ε, ατομικές, περιφερειακές και εθνικές δράσεις. Τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε τα όσα πετύχαμε. Η οικονομία της Ευρώπης δεν είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν, αλλά είναι μια ζωντανή πραγματικότητα είναι ε, ο ακρογωνιαίος λίθος, είναι τα, ο ιστός ας πούμε της ε, κοινωνίας μας. Είναι εύκολο να αισθανόμαστε ότι είναι δικό μας. Ε, αλλά δεν είναι για όλους έτσι. Θα πρέπει να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να εξερευνήσουν το παρελθόν τους, να δουν ποιοι είναι και πώς εντάσσονται στη σημερινή κοινωνία, ό,τι και αν έχουν ζήσει, ό,τι και αν έχουν περάσει. Είναι η δέσμευσή μας προς τους Ευρωπαίους και πιστεύω ότι όλοι Μαζί θα συνεχίσουμε προς αυτό το στόχο. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι η ομάδα μου δημιούργησε το δικό μας παιχνίδι για να θυμόμαστε αυτό το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, για να απαθανατήσουμε τη δουλειά που κάναμε το 18 και εσείς είσαστε οι πρώτοι που λαμβάνετε αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν το έχω λάβει καν, έχω, <laughs> αισθάνομαι πραγματικά προσβεβλημένη, αλλά το έφερα ε, για τα μέλη της Επιτροπής. Και φυσικά το πρώτο αντίτυπο ας πούμε, αυτού του παιχνιδιού πάει στην Πρόεδρο. Πέτρα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι για την τελευταία μας συνεδρίαση ε, θα λάβουμε και ένα δωράκι. Και είναι σημαντικό να ε, αντιληφθούμε ότι αυτοί οι οποίοι στην Επιτροπή εργάζονται με το ζήτημα ε, του, πολιτισμού πραγματικά ε, ενδιαφέρονται για αυτό και θέλουν να προωθήσουν τα πολιτισμικά ζητήματα, όμως ε, πολύ συχνά δεν εξαρτάται μονάχα από μια γενική διεύθυνση εάν θα ακολουθήσει ε, η επιτυχία, διότι υπάρχουν πολλοί άλλοι στην Επιτροπή, πολλοί άλλοι επίτροποι οι οποίοι έχουν και αυτή την άποψή τους ε, και εν τέλει ε, στο τέλος η μία ή η άλλη υποχρέωση φρενάρεται εν τέλει. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στους ε, μεμονωμένους εργαζομένους και αυτό ε, το οποίο προωθεί τελικά στο ε, πολιτικό της θεματολόγιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε και πάλι λοιπόν για το δώρο και τώρα θα ακολουθήσει η συζήτηση. Βλέποντας όμως το ρολόι θα σας καλούσα να περιοριστείτε στα δύο λεπτάκια. Η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλη την ομάδα σας. Γυναίκες ήσασταν κυρίως. Δουλέψατε με εντυπωσιακό τρόπο. Εντοπίσατε τρεις διαστάσεις. Αυτό που είχαμε ζητήσει. Μία ολοκληρωμένη διακυβέρνηση, διαχείριση, ε, όπου θα συμμετείχαν όλες οι γενικές διευθύνσεις με τρόπο ε, οριζόντιο. Νομίζω 14 ε, γάμα δέλτα συνεργάστηκαν ε, το θέμα της πλατφόρμας με τους stakeholders και η σχέση με το Κοινοβούλιο. Τρεις άξονες λοιπόν. Αυτό ήταν ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας και ελπίζω μια και αναφερθήκατε στο φόρουμ, ε, ελπίζω να διατηρήσετε αυτό το συντονισμό με τις άλλες γενικές διευθύνσεις και έναν έντονο διάλογο με, τις, ε, με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους stakeholders. Δεύτερο στοιχείο Δίκιο έχετε, Πρόεδρε. Θέλαμε ε, ε, ευρωπαϊκές εμπειρίες, ε, γιατί πάντα δεν ήταν έτσι. Τώρα έχουμε τις βάσεις με τα 10 θέματα που εντοπίσαμε. Κοινά ευρωπαϊκά θέματα και το διάλογο που ενεργοποιήθηκε. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποιες προτεραιότητες. Έχουμε τα, τους πέντε πυλώνες που αναφέρατε και έχουμε και αυτή την ομάδα εργασίας που θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη. Και έτσι θα πρέπει να προβάλλουμε ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή διάσταση των μεγάλων θεμάτων. Το σχέδιο δράσης το σχέδιο εργασίας δεν είναι μεγάλη πολιτική κατεύθυνση. Εμείς θέλαμε να διατηρηθεί αυτή η governance ε, που είχαμε το 18. Το σχέδιο εργασία είναι κάτι πολύ λιγότερο, ας πούμε. Ε, γιατί δεν θέλω να αποστρέψουμε το βλέμμα από τη σημαντική δουλειά που έγινε το 18. Ε, δύο πράγματα τώρα και κλείνω. Αυτά τα χρόνια στοιχηματίσαμε σε αυτήν την οριζόντια προσέγγιση. Ε, το βάλαμε και στο Εράσμους και στην ε, Δημιουργική Ευρώπη και προβλέψαμε και επιπλέον πόρους με, για την έρευνα, με την ε, συνεργασία για την ανάπτυξη. Είναι μια κοινή δουλειά. Στην Δημιουργική Ευρώπη υπάρχει μια νέα γραμμή για την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή η νέα γραμμή είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν αρκεί. Αυτό που μας ανησυχεί είναι τα λεφτά που προβλέπονται από την Κομισιόν ε, είναι 1,8 δις. Εμείς ζητήσαμε 2,4. Ε, αυτό εξαρτάται από την επόμενη διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να υπάρξει πίεση προς το Συμβούλιο για να συνενέσει να δώσει περισσότερα λεφτά. Και θα πρέπει να υπάρξει μια συγχώνευση όλων των πόρων όλων των πόρων από τα διάφορα προγράμματα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Διάκονου. Ο κύριος Διάκονου. Ευχαριστώ πολύ. υπέροχα. Νιώθω όπως όταν ήμουν ε, μαθητής ε, και στο τέλος της χρονιάς πάντοτε είχαμε μια ωραία ε, χρονιά αποφύτησης και κάπως έτσι είναι η ατμόσφαιρα και σήμερα, κάτι το οποίο με συγκινεί ιδιαίτερος. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να ευχαριστήσω αυτή την Επιτροπή, διότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε ασχοληθεί και συνεργαστεί στενά και αποτελεσματικά με διάφορα θέματα και στην συνέχεια ψηφίσαμε και ε, σημαντικά ε, έργα όπως ήταν για παράδειγμα το πολιτιστικό έτος. Ε, στις διαπραγματεύσεις όμως θα πρέπει να ομολογήσω ότι είχα την εντυπώση ότι το πιο δύσκολο ήταν πως εμείς ως κοινοβούλιο έπρεπε να πείσουμε ότι είμαστε εταίροι για όλη τη διάρκεια του έργου ήταν δύσκολο, όμως είναι απίστευτο το, το καταφέραμε και αυτό με την υποστήριξη της Επιτροπής και λιγότερο του Συμβουλίου. Και θα επιθυμούσα να παραμείνει ως έχει. Οι στρατηγικές ε, για την ε, συνέχιση των ε, προγραμμάτων θα πρέπει να εφαρμοστεί τώρα. Όμως, Επίσης είναι σημαντικό να προωθήσουμε αυτό το έργο και λυπάμαι εν μέρη που ε, δεν ε, θα συμμετάσχω σε άλλη μία θητεία στην Επιτροπή ε, Κουλτ. Όμως το σημαντικότερο είναι το τι θα προκύψει από, αυτά, από αυτό το πρόγραμμα, τι θα μας μείνει. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και πάλι την Επιτροπή για το ότι ε, ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτό και όλο αυτό δείχνει ότι ο πολιτισμός έχει αποκτήσει μια σημαντική θέση ε, στον ε, ευρωπαϊκό πολιτισμό, στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Ευχαριστώ πολύ για τον ενθουσιασμό που έχει δημιουργήσει ε, αυτό το έτος ε, ανάμεσά μας. Όμως ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία, πετύχαμε πολλά πράγματα και, το, και εν τέλει η Επιτροπή ήταν αυτή που μας βοήθησε περισσότερο και όχι τόσο το Συμβούλιο. Ήμουν εισηγητής μιας γνωμοδότησης όπου ασχοληθήκαμε σχετικά με την προώθηση των αξιών ε, και αυτό το οποίο μας λείπει λοιπόν είναι η προώθηση της ε, πολιτισμικής κληρονομιάς. Ε, δεν μιλάω όμως για μουσεία, για το Λούβρο, μιλάω για τα μικρότερα πραγματάκια, τα οποία όμως θα θεωρώ ότι θα χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Αυτό το οποίο επίσης θα ήθελα να σας πω είναι ε, οι ευχαριστίες που θα ήθελα να δώσω. Μιλάω τελευταία φορά εδώ. Ευχαριστώ την Πέτρα, ευχαριστώ την κυρία Κώστα. Διότι εσείς ήσασταν που ε, ηγηθήκατε πολύ καλά ε, μέσα στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ όσους μας υποστηρίξατε είχαμε τρομερή υποστήριξη. Ευχαριστώ όλους και όλες τις ε, συναδέλφους. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι ε, δεν ήταν χαμένος ο χρόνος μου σε αυτή την επιτροπή. Ασχοληθήκαμε με σημαντικά προβλήματα, με το, με το Erasmus+, με το Creative Europe, με το ε, πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες ε, και αυτή τη στιγμή όχι μόνο υπερασπιστήκαμε το Erasmus Plus αλλά το μεγαλώσαμε κιόλας. Ε, είχαμε τρομερές επιτυχίες και ευχαριστώ όλους για αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι σίγουρα αυτό που ενώνει τις γενιές μεταξύ τους. Και αυτό ισχύει και για ένα τραγουδάκι που τραγουδάει η μητέρα στο παιδί της, αλλά και στα εθνικά μας μνημεία. Και δεν υπάρχει πολιτιστική κληρονομιά χωρίς μετάδοση στις επόμενες γενιές. Είναι ζωντανή λοιπόν η πολιτιστική κληρονομιά και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να γίνουν ακόμα πιο προσβάσιμες αυτές οι σημαντικές αξίες. Θα ήθελα εδώ να χαιρετήσω την ε, σημαντική προσπάθεια που έγινε στη δική μου περιοχή, έτσι ώστε το κάστρο και η βιοτεχνία γύρω από το Λίνεβιλ να διατηρηθεί και να ξαναζήσει. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες πρωτοβουλίες, έξυπνο τουρισμό με νέα δίκτυα και τη νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων που δημιουργήθηκε. Πιστεύω πραγματικά ότι τα ιστορικά μνημεία, τα οποία θα πρέπει να αντισταθούν στα φυσικά φαινόμενα και στους σεισμούς, να υλοποιηθεί. Δεν ξέρω όμως και δεν κατάλαβα αν υπάρχει και ε, χρηματική στήριξη σε αυτή την πρωτοβουλία. Πρέπει να περιμένουμε ένα σεισμό στην Ελλάδα ή στην Ιταλία για να αποδεσμεύσουμε κάποια εκατομμύρια ευρώ. Όταν έπρεπε να σώσουμε το τραπεζικό σύστημα, πολύ περισσότερα χρήματα διατέθηκαν και αυτό αμέσως. Είναι λοιπόν λυπηρό που παραδείγματο χάρη το Κολυσσέο σήμερα ανακαινίζεται χάρη έναν ιδιωτικό χορηγό, την ε, εταιρεία TODS θα πρέπει ίσως να ξαναδούμε λίγο τις προτεραιότητές μας, τα μνημεία μας και τον πολιτισμό μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σόντροβα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα να βοηθήσω και να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την συνεργασία που είχαμε όσον αφορά αυτό το τελευταίο έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, συζητήσαμε για αυτήν την νέα πρωτοβουλία και αυτά τα 18.000 ε, γεγονότα, εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν, βοήθησαν ε, τις μικρές κοινότητες, ε, τους μεγάλους δήμους, τα κράτη να συμμετέσχουν σε αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια. Εμείς είδαμε στην Τσεχία τον πρόεδρο, αλλά και μικρές κοινότητες που συμμετείχαν σε αυτήν την πρωτοβουλία και παραδείγματος χάρη ο γνωστός διευθυντής ορχήστρας που ήρθε και μαζί με την ορχήστρα την Εθνική Ορχήστρα και γειτονικέ ε, περιφέρειες από την Πρατισλάβα, από την Κρακοβία, από το Πέρτ, οργάνωσαν μια μεγάλη εκδήλωση, καθώς και πολλές συζητήσεις, εκθέσεις, σύγχρονης τέχνης. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δημιουργικό πρόγραμμα με φωτογραφίες, με κινηματογραφικές ταινίες και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι είναι κρίμα αν όλη αυτή η δυναμική του 2018 δεν συνεχιστεί. Ακούσαμε αυτό που είπε ο κύριος Διάκονο. Εγώ ελπίζω πραγματικά το επόμενο Κοινοβούλιο, η επόμενη Επιτροπή θα συνεχίσει σε αυτήν την δυναμική με νέες πρωτοβουλίες και θα συνεχίσει αυτό που έγινε φέτος. Θα ήθελα και επειδή είναι ίσως η τελευταία φορά που βρίσκομαι εδώ να ευχαριστήσω όλους, ε, όλα τα μέλη της Επιτροπής και τους συνεργάτες μου. Ευχαριστώ πολύ, Julie Ward. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάναμε και ότι μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε όλους τους πολιτισμούς και όλες τις παραδόσεις που ζουν στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά δεν αποκλείει κανένα, ιδιαίτερα τον Ισλαμικό πολιτισμό. Υπάρχει ένα κίνημα στην Ευρώπη για να δαιμονοποιήσουμε το Ισλάμ. Πολλές από τις παραδόσεις μας ε, προέρχονται από τον Ισλαμικό πολιτισμό. Και βεβαίως εγώ συνεργάστηκα με πολλές πρωτοβουλίες και γιορτάσαμε τις Ισλαμικές παραδόσεις και όλα αυτά που έχει προσφέρει αυτός ο πολιτισμός στην επιστήμη, στην ιατρική, στην ε, αστρονομία, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς τι σημαίνει να είναι σήμερα κάποιος Ευρωπαίος. Και οργανώσαμε συγκεκριμένες εκθέσεις από τα Ευρωπαϊκά Μουσεία, τις Ευρωπαϊκές Συλλογές των Ευρωπαϊκών Μουσείων, που προέρχονται από την Ισλαμική παράδοση και τον Ισλαμικό πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση ακριβώς αυτό ε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια αποκλεισμού και άρνησης του Ισλαμικού στοιχείου από τον πολιτισμό μας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την ε, εβραϊκή παράδοση και μάλιστα ο Μάκο Μέλ, ο οποίος είναι επικεφαλής ε,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 είναι λίγο η σταχτομπούτα των ε, επιτροπών. Έγινε αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι είναι θετικά αυτά που τα υπογραμμίσουμε και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ στην Επιτροπή μας, στο Κοινοβούλιο, ε, δώσαμε μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα και ένα δεύτερο ότι έγινε μία συνεργασία. Ε, υπάρχει ένα θέμα όμως που αφορά τις κυβερνήσεις. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι τα αιτήματα που έχουμε υποβάλει, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και από εδώ και πέρα το λόγο έχουν οι κυβερνήσεις. Ε, επίσης, η διασύνδεση με το InvestEU ε, θέτει νέες προκλήσεις. Είναι μεγάλο θέμα αυτό και θα πρέπει να γίνει και ένας προβληματισμός για άλλα θέματα τα οποία έχουμε εντοπίσει αυτά τα πέντε χρόνια στα πλαίσια του θεματολογίου για τον πολιτισμό. Πρέπει όμως να αναλάβει τώρα το επόμενο κοινοβούλιο για να τα υλοποιήσει. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, ευχαριστώ τις γενικές διευθύνσεις με τις οποίες συνεργαστήκαμε για τη συνεργασία. Τώρα θα έχουμε μια νέα Επιτροπή Πολιτισμού, ε, η οποία ελπίζω να προωθήσει αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπετε ότι είναι εξαιρετικά αρμονική η σημερινή μας συνεδρίαση. Ήταν πάντα έτσι. Θα ήθελα τελειώνοντας να αναφερθώ σε ένα έγγραφο που αναφέρεται στην 9η Απριλίου, Digital Day, ψηφιακή ημέρα, που ουσιαστικά οργανώνεται στα κράτη-μέλη και προέρχεται από το DigiConnect κατά την άποψή μου. Έχετε επαφή, η δική σας γενική διεύθυνση έχει επαφή με αυτή την πρωτοβουλία, αυτή τη Γενική Διεύθυνση, γιατί έχω την εντύπωση ότι ξαφνικά τους ήρθε η ιδέα να προετοιμάσουν κάτι πολύ εσπευσμένα, κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για αυτήν την ημέρα την ψηφιακή και πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συμπεριλάβουμε και την πολιτιστική κληρονομιά σε αυτό. Δεν ξέρω, θα περίμενα κάτι λίγο πιο φιλόδοξο, λίγο πιο προετοιμασμένο, λίγο πιο... εμπειριστατωμένο. Έχω την εντύπωση ότι ξαφνικά θυμήθηκαν ότι 9 Απριλίου υπάρχει αυτή η ημερίδα και ξαφνικά θέλησαν να συμπεριλάβουν και άλλους τομείς. Έχω την εντύπωση όμως ότι με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα τα ψηφιακά εργαλεία είναι εξαιρετικά σημαντικά για την πολιτιστική κληρονομιά, για τη διατήρησή της, για τη μετάδοσή της. Ε, αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση και φυσικά θα πρέπει ενδεχομένως να αποκτήσει βαθιές ρίζες στα κράτη-μέλη και δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εννοείται ότι ο σημερινός μας πολιτισμός, ε, οι σημερινές πολιτιστικές προσπάθειες και ό,τι κάνουμε σήμερα θα είναι η πολιτιστική κληρονομιά του μέλλοντος. Ε, η μετάδοση λοιπόν από τις παλιότερες, τις νέες γενιές. Είναι καθοριστικό στοιχείο αυτό που πρέπει να στηρίξουμε. Κάνουμε λοιπόν μια έκκληση για το μέλλον. Θα σας δώσω το λόγο για να ολοκληρώσετε και μετά θα περάσουμε και στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας ε, τις προτάσεις σας και τα σχόλιά σας. Ε, θα το ξέρετε αυτό σίγουρα. Σχετικά με το τελευταίο ερώτημα της Προέδρου, ναι, οι ε, Γενικές διευθύνσει Connect και ΕΑΚ ε, συνεργάστηκαν ούτως ώστε να προετοιμάσουν ένα κείμενο το οποίο θα καλούσε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν μεταξύ του. Έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αποτελεί ε, ένα πρωτοβήμα, δεν είναι ένα μακροσκελό προετοιμασμένο έργο. Σίγουρα μπορούμε να γίνουμε πιο φιλόδοξοι και ε, πάντοτε ε, πιεζόμαστε να γίνουμε πιο ε, φιλόδοξοι. Σίγουρα θα συνεχίσετε να το κάνετε αυτό και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Θέλουμε λοιπόν να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν το ότι θα πρέπει να συνεργαστούν. Είναι λοιπόν ένα πρώτο βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. να είστε βέβαιοι ότι και η επόμενη Επιτροπή ε, Κουλτ θα πιέσει ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν μας λέτε εσείς ότι είναι καλό αυτό, τότε χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε που ήσασταν ε, σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ για την καλή συνεργασία των τελευταίων χρόνων και για αυτούς που θα ακολουθήσουν σίγουρα θα συνεχιστεί ή ε, τόση καλή συνεργασία. Και φυσικά και εσείς είστε προσκεκλημένοι στη συνέχεια να γιορτάσετε μαζί μας. Ούτως ώστε να αποχαιρετήσουμε όμορφα αυτήν την ε, θητεία. Θα με παρακάλεσαν να ε, σας ενημερώσω ότι είναι και η πρόεδρος της Οϊρόπα Νόστρα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ την ε, Οϊρόπα Νόστρα, ε, η οποία πραγματικά συνεισέφερε στην χρονιά, για την, στην πολιτιστική χρονιά. Και τώρα περνάμε στην γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα για το δικαιώματα και τις αξίες. Πιστεύω ότι και εδώ μπορούμε να περιμένουμε καλά αποτελέσματα. Η Επιτροπή μας το υπερασπίστηκε έντονα. Δεν ήταν τόσο εύκολο ε, κατά τις ε, διαπραγματεύσεις. Μερικές φορές ήταν δύσκολο να προωθήσουμε τα θέλω μας στην Ελίμπε που είχε, ήθελε τα, ε, είχε τους δικούς της στόχους. Παρ' όλα αυτά όμως ε, κάνουμε πολύ καλή δουλειά να υπερασπιστούμε τα ε, συμφέροντα της Επιτροπής Κούλτ. Ευχαριστώ. Είμαι η τελευταία που θα μιλήσει στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού. Ε, σας ευχαριστώ για τα λόγια σας. Όταν ξεκινάμε μια διαπραγμάτευση, ε, υπάρχει ένας δεδομένος συσχετισμός δυνάμεων. Αλλά όλα πήγαν καλά. Οι διαπραγματεύσει ε, είχαν μια κάποια ένταση με την Επιτροπή, η οποία και το Συμβούλιο, που δεν είναι κατά ανάγκη στο γεωμικό σχήμα, δεν έχουν την ίδια άποψη κατά ανάγκη με εμά. Οι δύο άλλοι εταίροι μας επέτρεψαν να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Μετά από τέσσερι τριμερεί διαλόγους βρήκαμε μια μερική συμφωνία αρχέ Μαρτίου και το πρόγραμμα για το οποίο μιλάμε θα λέγεται ε, πολίτες, ε, ισότητα, δικαιώματα και αξίες. Έχουμε λόγους να είμαστε ικανοποιημένοι, θα τα πω όλα τους λόγους. Ε, δύο-τρεις θα αναφέρω μόνο. Καταρχάς το Συμβούλιο συμφώνησε τελικά για μια νέα πτυχή για την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό είναι ο τέταρτος στόχος του προγράμματος, αλλά διατηρήσαμε το δικό μας ε, στόχο για την ε, συμμετοχή των πολιτών. Ε, ήταν πολύ σημαντικό να μην υποχωρήσουμε εκεί. Και δεν υποχωρήσαμε. Το παλιό πρόγραμμα Ευρώπη των πολιτών διατηρείται μέσω των στόχων των γενικών με μια καλύτερη ισορροπία στο τελικό κείμενο από αυτό που υπερασπιζόταν η Επιτροπή Ελευθεριών, η ΛΥΜΠΕ και σε ένα άλλο άρθρο, το οποίο συμφωνήθηκε στον τρίτο τρίμιο, τρίλογο, όχι τέταρτο, για την συμμετοχή και δέσμευση των πολιτών θα έχουμε τρεις ε, πτυχές, ό,τι, αφορούν, ό,τι αφορά τη μνήμη. Ε, κάναμε, είχαμε πρόβλημα λιγάκι με το θέμα αυτό της μνήμης. Ε, το η δεύτερη πτυχή αφορά τη δημοκρατική συμμετοχή και η τρίτη πτυχή αφορά την δημοποίηση και το δίκτυο των πόλεων ε, αδελφοποίηση μάλλον και δίκτυο πόλεων. Ε, ε όσοι συναντάνε τοπικές οργανώσεις όπως εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι θα ενδιαφέρονται πάρα πολύ γι' αυτό. Θα δοθεί μια τελευταία μάχη, έτσι, εμείς γενικώ και ορίστος. Τέλος ε, το Κοινοβούλιο θα δώσει μια ακόμα μάχη που θα είναι η μάχη του προπολογισμού, γιατί η συμφωνία είναι μόνο προσωρινή και οι δημοσιονομικές πτυχές ε, εξαρτώνται από τις οριζόντιες διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για το επόμενο πουδουπού, το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. υπενθυμίσω ότι για αυτό το ε, κομμάτι θέλουμε τριπλασιασμό του προϋπολογισμού, 500 εκατομμύρια δηλαδή, για το δικό μας κομμάτι. Ελπίζω ότι οι μελλοντικοί συνάδελφοι θα έχουν την ίδια επιμονή και μαχητικότητα με εμά. Στι 17 Απριλίου στο Στρασβούργο, στην Ολομέλη, θα γίνει τελική ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σου και ευχαριστώ που ε, υπερεσπίστηκες ισχυρά τις ε, θέσεις της Επιτροπής μας. Ομολογώ ότι θα ε, προτιμούσα να ακολουθούμε τη διαδικασία που κάναμε με τα δικά μας ε, προγράμματα, πρώτη αναγνώση στην Ολομέλεια και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι συζητήσεις. Εδώ έχουμε ε, ένα αποτέλεσμα όπου δεν ξέρουμε πόσα χρήματα θα είναι διαθέσιμα εν τέλει. Όμως ε, βασίζομαι στο επόμενο κοινοβούλιο και την επόμενη επιτροπή η οποία θα συμμετάσχει στη διαδικασία ότι θα υπερασπιστεί ούτως ώστε το σχέδιο που θα προκύψει να είναι έτσι όπως το επιθυμούμε. Δεν ήταν στο χέρι μας διότι η Βασική Επιτροπή ήταν η ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστούμε όμως και πάλι για το έργο που έχεις ε, κάνει και η Ζαμπίνε Φεράιν και η κυρία Κώστα ζήτησαν το λόγο. Έχω ένα ερώτημα στο πρόγραμμα Ευρώπη για τους ε, πολίτες, εκεί όπου ε, το ζήτημα αφορά τις ε, εταιρικές σχέσεις μεταξύ των πόλεων, πώς είναι η κατάσταση σχετικά με την πρόσβαση στο πρόγραμμα για μικρές οργανώσεις, μικρές εταιρικές σχέσεις. Αυτό ήταν πάντοτε ένα σημαντικό θέμα της Επιτροπής, όμως η δική μας Επιτροπή πάντοτε ε, ήθελε και μικρότερες ομάδες να έχουν τη δυνατότητα ε, να ε, δημιουργούν αυτές τις εταιρικέ σχέσεις, μικρότερες πόλεις, μικρότερες κοινωνίες. Υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κώστα. Ευχαριστώ τη Σιλβή για τη δουλειά της. Χαίρομαι που μπήκε η λέξη όχι ηθαγένεια, αλλά πολίτες στον τίτλο πολίτες, λυπάμαι, και ξέρω βέβαια τι έδωσε μάχη, λυπάμαι που δεν υπάρχει ε, η αναφορά δραστηριότητα για την εκπαίδευση των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του προγράμματος, ε, υπήρχε στο Εράσμους, αλλά τέλος πάντων. Ε, καταγράφω όλα τα σημαντικά πράγματα που πέτυχες και ελπίζω ότι η δέσμευση για την αύξηση του, της δικής μας γραμμής του προϋπολογισμού να υλοποιηθεί. Γιατί ο κίνδυνος είναι να χάσουμε στο συνολικό πρόγραμμα, στο merging program, την ιδιαιτερότητά μας. Έδωσες μάχη μου; γι' αυτό και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Σιλβί. Ναι, θέλω να ξεκαθησυχάσω, Σιλβία. Είναι όλα τα μικρά αυτά σχέδια συμπεριλαμβάνονται. Ωραία. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν και με μεγάλη εμπιστοσύνη αναποθέτουμε όλα αυτά στην επόμενη επιτροπή, στην επόμενη επιτροπή πολιτισμού, στην επόμενη πολιτι... επιτροπή ΛΥΜΠΕ και νομίζω ότι φτάνουμε στο τελευταίο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι τα διάφορα. Η Τζούλη έχει το λόγο. Θα ήθελα να αναφερθώ στα σχέδια για το 2019. Εγώ μιλούσα στην Πρατισλάβα την Παρασκευή σε ένα συνέδριο και υπήρχε κάποιος εκεί ο οποίος συμμετείχε στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων. Και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές επιθέσεις ε, το ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται στον καλλιτεχνικό διευθυντή και σε καλλιτέχνες γιατί συμμετέχουν στον προγραμματισμό στο Plovdiv και μάλιστα έχω εδώ μια ολόκληρη έκθεση, πολλές σελίδε που αναφέρεται σε όλες αυτές τις επιθέσεις κατά των ε, καλλιτεχνών και αυτό βεβαίως από μέρους ακροδεξιών δυνάμεων, επιθέσεις και κατά πολιτικών. Και πραγματικά θα ήθελα να δραστηριοποιηθούμε σαν Επιτροπή, γιατί εδώ πρόκειται για την ακαιρεότητα του προγράμματος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζουμε, χρηματοδοτούμε και πρόκειται για θεμελιώδεις αξίες και θα πρέπει με μεγάλη σαφήνεια να μιλήσουμε για αυτές τις επιθέσεις. Υπήρξαν διαμαρτυρίες τις τελευταίες μέρες, συγκεκριμένα μέχρι και το Σάββατο και υπήρξε ε, συγκεκριμένη διαδήλωση κατά του καλλιτεχνικού διευθυντή ζητούσαν την ε, παρέτησή του. Και γιατί, διότι υπήρχε μια ομάδα καλλιτεχνών ΛΟΑΔ αυτή τη στιγμή οτιδήποτε δεν είναι παραδοσιακό ή δεν εκπροσωπεί τα δύο φύλλα με ξεκάθαρο τρόπο, είναι αντικείμενο επιθέσεων. Πρέπει να αντισταθούμε, πρέπει να προσπίσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Και μάλιστα πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε μια αντιπροσωπεία και κάτι να πούμε. Δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας λέγοντας ότι όλα πάνε καλά πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα συμβαίνουν στην πόλη αυτή και θέλω πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι της Επιτροπής μας να διαβάσουν αυτή την έκθεση και να δραστηριοποιηθούμε, να σχολιάσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ Τζούλη για αυτήν την ενημέρωση. Για μας είναι κάτι καινούριο, η Χέλγα. Εγώ ήμουν ε, η επικεφαλής της αντιπροσωπείας στο Πλόπτικ και η Τζούλη και άλλοι συμμετείχαν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν υπάρχει ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για τον πολιτισμό, τέτοιου είδους φαινόμενα πολλές φορές εμφανίζονται και θα είμαι πολύ, αν θέλετε, ειλικρινής ε, για το θέμα αυτό. Υπήρξε μια έκθεση που αφορούσε τον Χόνεκερ, που αφορούσε το τείχος του Βερολίνου και δεν ξέρω αν οι επιθέσεις ήταν ε, ε τεκμηριωμένες ή όχι. Σίγουρα πρέπει να εξετάσουμε την περίπτωση, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αν είναι ακροδεξοί ή όχι αυτοί που επιτίθενται Πρέπει να ενημερωθούμε, αυτό λέω, πρέπει να μιλήσουμε και με αυτούς που επιτίθενται, πρέπει να ε, αναφερθούμε και στον καλλιτεχνικό διευθυντή. Ε, έχετε φέρει αυτή την έκθεση, αλλά πρέπει πρώτα να τη διαβάσουμε. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ αυτό θα πρότεινα, ότι πρέπει να το εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή, να έχουμε επαφές ε, επιτόπου και η γραμματεία της Επιτροπής θα επιληφθεί του θέματος αυτού και θα επανέλθουμε όταν έχουμε πιο συγκεκριμένη ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζούλη. Και τώρα το πραγματικά τελευταίο τελευταίο σημείο. Έχετε κάτι να προσθέσετε στα διάφορα, όχι. Στο τέλος αυτής της νομοθετικής περίοδου στο τέλος της θητείας αυτής της Επιτροπής. Νομίζω ότι πολλοί πήραν το λόγο και είπανε είναι η τελευταία φορά που παίρνω το λόγο, είναι η τελευταία φορά που αναφέρομαι σε θέματα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ολοκληρώσαμε τη θητεία μας. Ήταν για μένα μεγάλη τιμή που μπόρεσα να προεδρεύσω αυτή της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Συνεργαστήκαμε με τόσο πολλούς που πραγματικά έχουν δεσμευτεί για θέματα που αφορούν ε, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τους νέους, και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την προκάτοχό μου στο πρώτο μισό αυτής της θητείας, τη Σίλβια Κώστα, η οποία με μεγάλη επιτυχία προώθησε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, έτσι ώστε να αποκτήσουν τη σημασία που τους αξίζει στην ευρωπαϊκή πολιτική τα θέματα αυτά. Δεν ήταν εύκολη η δουλειά μας και στο τέλος της θητείας μας Ελπίζω να βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι τα θέματα αυτά έχουν αποκτήσει τη σημασία που τους αξίζει, αλλά ελπίζω ότι η εργασία όλων μας, η εργασία της προκατόχου μου, της Σίλβια, με τις ίδιες πολιτικές προτεραιότητες, να βελτιώσαμε λίγο τα πράγματα στο τέλος αυτής της θητείας. Βεβαίως Ξέρουμε τι σημασία δίνει και η Επιτροπή στα θέματα αυτά και ελπίζω κάποια στιγμή να μπει στην καρδιά και όχι στο τέλος ε, των πολιτικών προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής πολιτικής ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Συνεχίσαμε τις ε, μάχες και τις προσπάθειές μας και πιστεύω ότι σήμερα στην Ευρώπη έχουν όλοι καταλάβει ότι χωρίς μία δέσμευση στον τομέα του πολιτισμού και της ε, παιδείας δεν μπορεί η Ευρώπη να συνυπάρξει. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν τα κράτη στο εσωτερικό αυτής της Ευρώπης. Μιλάμε για την πολιτιστική κληρονομιά, για όλα τα επιτεύγματά μας και πραγματικά διαπιστώσαμε ότι με τέτοιες πρωτοβουλίες τα κράτη-μέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Τελικά πετύχαμε να πείσουμε τους πάντες ότι αυτή η πρωτοβουλία άξιζε τον κόπο και αυτό που κάναμε φέτος ήταν πολύ σημαντικό για το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σαν συντονιστές, ιδιαίτερα τη Χέλγα που έχει και αρμοδιότητες σε θέματα δημοσιονομικά. Ευχαριστώ πολύ για όλη σας την στήριξη γιατί πραγματικά η στήριξη και η αύξηση των κονδυλίων για προγράμματα πιλωτικά και μη στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα. Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και στις επόμενες θητείες. Στηρίζουμε την δημιουργία, στηρίζουμε τον πολιτισμό, στηρίζουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα αναφερθώ εδώ στη σημαντική οδηγία που τελικά καταφέραμε μετά από πολλές προσπάθειες και αγώνες ε, να περάσουμε με νομίζω ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το θέμα του νέου σώματος αλληλεγγύης, ένα άλλο σημείο που μας απασχόλησε και τα δύο μελλοντικά προγράμματα Creative Europe και Erasmus Plus. Νομίζω και για τα δύο αυτά προγράμματα έχουμε συνεισφέρει έτσι ώστε το μέλλον να αποδείξει και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επόμενη Επιτροπή Πολιτισμού να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες αυτές. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν θα επανεκλεγώ και θα είμαι παρούσα στην επόμενη θητεία, θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου και όσον αφορά τη συνέχεια αυτών των προγραμμάτων, αλλά και όσον αφορά την στήριξή τους. Εκθέσεις πρωτοβουλίες, ακροάσεις, ε, εργαστήρια, workshop, ιδέες και πρωτοβουλίες που μπορέσαμε να στηρίξουμε σε θέματα όπως η κατάρτιση, η δημιουργία, ο αθλητισμός, ε, οι ψηφιακές δεξιότητες, η κατάρτιση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής μας, όλους τους συνεργάτες, τους βοηθούς, τις βοηθούς, ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου, τη γραμματεία της Επιτροπής μας, τους διερμηνείς και τις διερμηνείς, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να εργαστούμε, τους εκπροσώπους ε, του Συμβουλίου, της Επιτροπής Περιφερειών, τους εκπροσώπους των ε, εθνικών φορέων και οργανισμών, των διεθνών οργανισμών που με την εμπειρογνωμοσύνη τους και τις γνώσεις τους μας στήριξαν τα τελευταία χρόνια. Και αυτά που πετύχαμε και αυτά που δεν πετύχαμε Έχουμε μπροστά μας τις ε, εκλογές και νομίζω ότι πολλές ιδέες και πολλές μελλοντικέ πρωτοβουλίες θα συνεχίσουν να μας εμπνέουν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους γιατί πιστεύω ότι η προσπάθειά μας ήταν συλλογική. Τα αποτελέσματα για τα οποία είμαστε περήφανοι είναι συλλογικά. Ήταν εξαιρετική συνεργασία μαζί σας τα τελευταία χρόνια δεν συμφωνούσαμε πάντα, αλλά είναι και τόσο βαρετό να συμφωνείς πάντα με όλους. Νομίζω ότι μέσα από την αντιπαράθεση και τη συζήτηση βγήκε κάτι θετικό και θεωρώ επίσης ότι αυτό αποδείχτηκε από τα αποτελέσματα με ένα πολύ φιλικό και συλλογικό τρόπο μπορέσαμε να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας για να στηρίξουμε τον πολιτισμό και όλους τους τομείς για τους οποίους έχουμε αρμοδιότητα. Θα ήθελα να σε ευχηθώ σε όλους κάθε καλό. Είτε είστε εδώ στο Κοινοβούλιο, είτε είστε κάπου αλλού. Σας εύχομαι κάθε καλό, επιτυχία για αυτούς που θα επανέλθουν εδώ, για αυτούς που είναι υποψήφοι και για αυτούς που δεν είναι. Όπου και να είστε, Ελπίζω να παραμείνετε δεσμευμένοι και πιστοί στην ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που αφορά τον πολιτισμό. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Η Σαμπίνε. Αυτή είναι η ε, πρώτη συνεδρίαση την οποία δεν ολοκληρώνω εγκαίρως ε, και θα πρέπει να συμβεί αυτό διότι Συμφωνώ απολύτω ε, με τις ευχαριστίες ε, που έχεις δώσει. Δεν θα ε, ευχαριστήσω όλους όσους ανέφερες, διότι ο κατάλογος είναι μεγάλος. Πιστεύω όμως ότι αυτό το οποίο λείπει από τις ευχαριστίες σου και το οποίο ξεχνάμε είναι ευχαριστίες σε σένα. Ευχαριστούμε την Σίλβια επίσης για το πρώτο μισό ε, πιστεύω ότι ε, χάρη στην ηγεσία σας καταφέραμε πάρα πολλά, μεταξύ άλλων και την προσοχή η προσοχή σε άλλες επιτροπές. Θυμάμαι για παράδειγμα ε, την Ήτρε, έχουμε την Επιτροπή Βιομηχανίας, ε, και εκεί ακόμα ε, μπορέσαμε να ε, επηρεάσουμε, καταφέραμε πολλά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό οφείλεται χάρη στην στενή και καλή συνεργασία εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά και το αγωνιστικό τρόπο με τον οποίο όλοι, αλλά και εσύ, προώθησες και προωθήσαμε τον πολιτισμό σε άλλους συναδέλφους και σε άλλες επιτροπές. Ήταν αναγκαίο μερικές φορές ε, με αποφασιστικότητα και σκληρότητα να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, συναδέλφους και τους ε, συντονιστές ακόμα και αν υπήρξαν διαφωνίες βρήκαμε έναν πολύ καλό δρόμο προς τα εμπρός. Ευχαριστώ πολύ Πέτρα και πιστεύω ότι μαζί μου συμφωνούν και όλοι οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ. Χέλγα από πλευράς μου. Ευχαριστώ ε, Πέτρα αλλά και την ε, Σίλβια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας. Δεν θα ε, είμαι υποψήφια και πάλι. Είναι προσωπική μου απόφαση Πάντοτε ήταν μεγάλη μου ευχαρίστηση και πάντοτε ήθελα να συμμετάσχω σε αυτήν την Επιτροπή, στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Ήταν ένας καλός συνδυασμός με την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών. Ε, αρχικά όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, το προσωπικό τους διερμηνείς, το προσωπικό μου Φριδερίκα Όλγα Μπένιαμιν, διότι ήταν ομαδική εργασία, υπήρχαν διαφωνίες φυσικά, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό σε ένα δημοκρατικό κοινοβούλιο, όμως ε, για χάρη του πολιτισμού και της παιδείας ήμασταν ενωμένοι και ήταν μεγάλη ικανοποίηση που συνεργαστήκαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σίλβια. Generosamente ricordato. Ευχαριστώ όλου, σας ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ και για αυτό το δεύτερο κομμάτι ε, υπό τη δική σου αιγίδα. Ε, ήταν πολλά τα σημαντικά θέματα, η στρατηγική για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, για τα, για τα ψηφιακά, αλλά βρήκαμε πάντα ένα σημείο ισορροπίας. Και εγώ έκανα μία επιλογή όταν μπήκα στην Επιτροπή Πολιτισμού για δεύτερη φορά, γιατί θεωρώ ότι η η αφιέρωσή μας και το όραμά μας, γιατί εγώ διεκδικώ το όραμα για αυτή την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό ευχαριστώ όλη την ομάδα του Νίλς ε, και όλο το προσωπικό για την βοήθεια. Μαζί με τους συντονιστές προσπαθήσαμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε να εξηγήσουμε ότι η κουλτούρα δεν είναι ένα κομματάκι, ας πούμε, αλλά μπαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, γιατί χωρίς μια πολιτιστική εκπαιδευτική και αλληλέγγυα θεώρηση και μία ενεργή ηθαγένεια δεν υπάρχει οικοδόμης Ευρώπης. Αυτή ήταν ε, η έννοια της δικής μας μάχης. Όχι μόνο να διεκδικήσουμε κάποια προγράμματα δηλαδή, αλλά να αποκαταστήσουμε στην πολιτική τον πολιτισμό. Έτσι. Σήμερα τα πράγματα αυτά είναι πιο ξεκάθαρα, χάρη και στην ε, οριζόντια προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Έτους Κοινωνίας, για το οποίο ευχαριστώ και την ε, Κομισιόν, και χάρη στη δική μας αφοσίωση ε, εξετάσαμε λιγάκι και τους ε, ευρωπαϊκούς κανόνες και το, και το ευρωπαϊκό μοντέλο, το οποίο πρέπει να επεκταθεί και στον ψηφιακό κλάδο. Σας ευχαριστώ ε, και τους εισηγητές και ευχαριστώ τη, τη συνεργασία με τις άλλες επιτροπές. Όλη αυτή η συνεργασία με τους συντονιστές και με τις άλλες ε, επιτροπές μας βοήθησαν να έχουμε μία πιο συνολική, ας πούμε, θεώρησα θεώρηση. Ε, όλα τα ταλέντα εδώ τα αξιοποίησαμε. Νομίζω ότι όλοι ικανοποιήθηκαν σε κάποιο βαθμό. Ε, βεβαίως, ε, αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε και μία από τις πιο ολιγάριθμες επιτροπές, αλλά έχει και το καλό του αυτό. Σας ευχαριστώ όλους για την συνεισφορά σας. Ευχαριστεί η ομιλήτρια και τους διερμηνείς ε, που έδωσαν και μάχη για την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια. Ε, σήμερα πρέπει να δώσουμε νέα προτεραιότητα σε νέα θέματα. Αυτά για την επόμενη Επιτροπή Πολιτισμού. Η επόμενη πολιτική... Επιτροπή Πολιτισμού θα έχει μια σημαντική κληρονομιά που πρέπει να τιμήσει. Και με καινοτομίε, αλλά χρησιμοποιώντας και αυτή τη στρατηγική που εμείς διαμορφώσαμε. Σας ευχαριστώ όλους, γιατί χωρίς ε, εσάς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τόσο συνολική δουλειά και για το καλό των πολιτών. Εγώ θα είμαι πάντα στο πλευρό όποιου πολεμάει στην Ευρώπη για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευση, την αλληλεγγύη και την ηθαγένεια. Και αν δεν με ξαναδείτε θα έχουμε άλλους τρόπους να βρεθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη συνεδρία και τώρα μπορούμε να βρεθούμε για ένα μικρό ποτάκι. Συγγνώμη. Silvia. μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σκιώδη επιτροπή. Αυτοί που δεν θα επανεκλεδούν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια σκιώδη επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ.